It's 10.30 and we need to start. Είναι 10 και μισή ώρα και θα πρέπει να αρχίσουμε. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλή δουλειά, διότι όπως θα θυμάστε αποφασίσαμε να ε, τα βάλουμε όλα την ίδια μέρα, να τα στριμώξουμε για να μην έχουμε αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής. Έγκριση της, ε, σχεδίου ημερήσιας διάταξης που δεν έχετε δει, μπορούμε να την εγκρίνουμε. And then I have a few και έχω μερικές ανακοινώσεις να σας κάνω. Όπως θα θυμάστε, σήμερα έχουμε κοινή, ακρόαση, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, ΑΦΚΟ Συνταγματικών Υποθέσεων. Οπότε στις 12 παρατέταρτο θα σταματήσει η συνεδρίαση για να συμμετέχουμε εκεί. Και οι διερμηνείς σας ενημερώνω ότι βρισκόμαστε στην 37η μέρα των κινητοποιήσεών μας ε, μετά από την εργασία τη διαμάχη που έχουμε με την ε, διοίκηση και δεν θα παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου. Συνεχίζει η πρόεδρο. Ε, συνεδριάζουμε με την Επιτροπή ΑΦΚΟ στον πέμπτο όροφο. Πάρτε το σανσέ. Θα έρθει η διαμεσολαβήτρια και ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ε, όπως πάντα αλλά ένα λόγο παραπάνω σήμερα. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι η Ίνα Σοκόλσκα, υπάλληλό μα, θα πάει στο Policy Department C ε, από τις 16 Ιουλίου. Παρευρίσκεται. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και ε, είναι καλή συνέχεια και καλή τύχη στο μέλλον. Και σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά στη γραμματεία. Καλά, δεν πάτε και πολύ μακριά. Θα τα ξαναπούμε. Θα σας ξαναδούμε. Και πολλές φορές πρώην υπάλληλοι μας ξανάρχονται για να μας βλέπουν. Όποτε θέλετε θα χαρούμε να σας βλέπουμε. Βεβαίω να εγκρίνουμε και τα πρακτικά πρέπει. Τις 16 Μαΐου που έχουν κυκλοφορήσει. Μπορούμε να, τις ε, να τα θεωρήσουμε εγκεκριμένα. Ωραία, ευχαριστώ. Στα διάφορα δεν έχω διάφορα. Ούτε ζήτησε κανείς συνάδελφος το λόγο. Προχωρούμε. Ψηφοφορία. Πολύ σύντομα η Ελεονόρα Εύη ζήτησε το λόγο παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Η αύξηση του προπολογισμού που προτείνεται για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή έχει ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου αυτού του διαμεσολαβητή στην, στην εκτέλεση των βασικών του καθηκόντων που είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η σωστή διοίκηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπήρξε μια σημαντική αύξηση καταγγελιών ατομικών όσο και περίπλοκων καταγγελιών που συνεχίζει να ε, να παρουσιάζει αύξηση και το 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβήτη μέσω των διαφόρων έρευνων και για τον ε, ε, Επίσης μεγαλύτερη ε, προστασία για τους ε, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Γίναν ε, δεκτές ειδικέ τα δικά μας αιτήματα μόνο μερικώς. Η αύξηση στον προπολογισμό θα ανταποκριθεί λοιπόν στις ανάγκες αύξησης του προσωπικού ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβήτη, βελτιώνοντας έτσι την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Νομίζω καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Βλέπω πως έχετε όλοι φέρει τις κάρτες σας, γι' αυτό άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now closed. And you see that it has been adopted. Thank you very much. And let's move now to the first petition. Και περνάμε στην πρώτη αναφορά που έχουμε για σήμερα. Είναι η 586 για την ε, Ε, για τα απόβλητα είναι σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Γαλλικίας. Έχουμε το κείμενο, είχαμε το κείμενο στα ε, γαλλικιανά, όχι στα ισπανικά. Ήταν λίγο περίπλοκο λοιπόν και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής που είναι ο κύριος Δίας Ντελκαστίγιο. Good Um, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Θα ήθελα να πω τα εξή για αυτή την αναφορά. Σε προηγούμενα ε, ανακοινωθένη η Κομισιόν ε, είπε ότι το περιφερειακό ε, πλάνο διαχείρισης των αποβλήτων της, της Γαλλικίας που υιοθετήθηκε στο 2011 αξιολογήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και βρέθη σύμμορφο προς την οδηγία ε, πλαίσιο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες ε, δράσεις ε, και μέσα για την επίτευξη των στόχων και έχει κατανεμηθεί ο προπολογισμό ε, με, ε, με λεπτομέρειες και με συγκεκριμένες πληροφορίες για τα συστήματα συλλογής, ε, συγκομιδής των, ε, ε αποκομιδή συγγνώμη, των αποβλήτων. Ε, υπάρχει δε και χώρο ταφή ε, πολύ ψηλό ποσοστό αποβλήτων πηγαίνει εκεί, το 2009 53%, ενώ πολύ λιγοστή ανακύκλωση γίνεται στη του 10%. Αναμένουμε οι τοπικές αρχές, αν δεν έχουν ήδη, ε, το έχουν ήδη κάνει, να ξεκινήσουν αξιολόγηση του πλάνου και να τροποποιήσουν όπως, ε, όπου δει και όπως δει και ε, η Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία μεταξύ τροποποιήθηκε ε, και έχουν εισαχθεί ψηλοί στόχοι ανακύκλωση και στόχος μείωσης των αποβλήτων που πηγαίνουν στις χωματερέ και συλλογή βιοαποβλήτων ε, μεταξύ άλλων ε, απαιτήσεων. Για τον λόγο αυτό, από τα μέσα του 2020 αναμένουμε την αξιολόγηση όχι μόνο για τη Γαλλική αλλά για όλα τα κρατημέλη να έχουμε πιο αυστηρά ε, σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Να θυμίσω ότι όταν μιλάμε για στόχους αυτή είναι επί τη βάση κράτους και όχι περιφέρεια σαν και αναμένουμε οι περιφέρειες της Ισπανίας και των υπόλοιπων χωρών της Ένωσης να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η Επιτροπή επίσης δεν μπορεί να αναμειχθεί στην επιλογή των μοντέλων διαχείρισης αποβλήτων. Είναι ένα θέμα που ε, εναπόκειται στις τοπικές αρχές. Και τέλος, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο που ξεκινά το 2021 για το Ταμείο Συνοχής, για παράδειγμα, η Κομισιόν δεν θα συγχρηματοδοτήσει μεχανικά και συγκαταστάσεις, ε, αποτεφρωτές και ηχοματερές πια. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση στην Ισπανία και όχι μόνο στη Γαλλικία χρειάζεται μεγάλη βελτίωση ε, για να ανακυκλωθεί πεθαίνονται περισσότερα παύλητα και να πηγαίνουν στις χωματερές λιγότερα. Ε, το 2016 η Ισπανία ε, ολόκληρη είχε ένα μέσο όρο 30% ανακύκλωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ισπανία μπορεί να μην καταφέρει να επιτύχει το στόχο του 2020 και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ξεκινήσει αυτό που λέμε το μηχανισμό ε, πρόορηση ή έγκυρη προειδοποίησης που είναι κομμάτι της κοινοτικής νομοθεσίας και που συνίσταται στο να έρθουμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό έχει ήδη γίνει την, την Άνοιξη φέτος και να προγραμματίσουμε δράσεις και μέτρα για τα επόμενα δύο χρόνια για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο σε, με τις, και να είμαστε σύμμορφοι με τις προθεσμίες. Έχουμε φτιάξει έναν οδικό χάρτη μάλιστα για την Ισπανία που περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και μέσα, δεν θα μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες, Πάντως εν γέννη το υπάρχον ε, ε, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την Γαλλική είναι σύμμορφο με τη νέα νομοθεσία και αναμένουμε αυτό το σχέδιο να αξιολογηθεί ε, συντόμως. Είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε το νέο σχέδιο μόλις το λάβουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε στο 1,5 λεπτό έκαστος. Ε, κυρία Σέντρα Ροντρίγκη. Okay. So the floor... Παρέμβαση εκτό μικροφώνου. Yes. Ε, Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω στου διερμηνείς δύο λόγια καταρχά. Γιατί έχουμε και διερμηνέα από την πόλη του Βίγο ε, συμπαράσταση για την απεργία τους. Δεύτερο, ε, στην πλατφόρμα κατά της εγκατάστασης αποτέφρωσης, η πλατφόρμα της Γαλλικίας κατά της αποτέφρωσης και υπέρ της ανακύκλωσης. Το 2013 έγινε αυτή η καταγγελία και ε, συμμετείχα και εγώ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι ήμουνα σε επαφή με τα μέλη της πρωτοβουλίας όλο αυτό το διάστημα και εξ ονόματος των Πρασίνων και της ε, Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας θέλουμε αυτή η αναφορά να εκπαιρεωθεί. Δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσαν να έρθουν ε, οι ε, αναφέροντες. Ε, θα πρέπει να παραμείνει όμως ανοιχτή αναφορά για διάφορους λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για αξιολόγηση και οι ίδιες αρμοδιότητες. Αυτές όμως μπορεί να παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Νόμο όπως και κάνουν. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει ε, ε, αυτό το θέμα των αποβλήτων και δεν ε, σέβεται την ιεραρχία των αποβλήτων γιατί δεν κάνει το διαχωρισμό των αποβλήτων για την ανακύκλωση. Άρα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα που προλαμβάνουν την παραγωγή αποβλήτων στην πηγή με το διαχωρισμό τους. Τι κάνει λοιπόν το κράτος τελικά, ή τα καίει τα σκουπίδια ή τα θάβει. 8 ε, χρόνια σιωπής και ε, Σογκάμα το 2017 δημοσίευσε η εταιρεία τα πεπραγμένα το 2015. 3,32 ε, τόνοι στους 100 να κυκλώνονται. Όλο και λιγότερα απόβλητα. Και μετά τι βλέπουμε μετά από 24 χρόνια λειτουργία του οργανισμού ανακύκλωση, η ε, κυβέρνηση τη Γαλλικία και η εταιρεία Σοκάμα δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης διακόπτη πρόεδρο. 1,5 λεπτό σα έδωσα Κοιτάξτε, περιμένω 4 χρόνια για αυτή την αναφορά. Ε, γιατί περιέργω και ε, είχε εξαφανιστεί. Ε, εξ των δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο εξ ονόματος των αναφέροντων, γιατί δεν του εκπροσωπείτε. Ναι, αλλά πρέπει να σας εξηγήσω τι γίνεται. Πρέπει να ακούσουμε και άλλους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Ναι, αλλά είμαι μέλος της Επιτροπής και ήμουν αρμόδια. there uh, are other members. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα αυτά που είπε η Κομισιόν ήδη τον Ιούλιο του 2015, πριν από τρία χρόνια δηλαδή. Και ακούσαμε επανάληψη της θέσεως. Ε, στόχοι επιτεύχθησαν σε εθνικό, όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων ε, στην Γαλλική, ε, άρα πρέπει να κλείσει το θέμα. Ναι, μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν το θέμα αυτό για να κάνουν εκστρατεία, αλλά δεν είναι εδώ η Επιτροπή Αναφορών βήμα και φόρουμ για προεκλογικές διεκδικήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σεντεροδρίγες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Νομίζω ότι είναι εκτός τόπου ε, να κατηγορούμε κάποιος ότι κάνει εκστρατεία όταν έχουμε τόσο σοβαρά ζητήματα στην ε, Γαλλικία. Δεύτερον, να πω ότι ε, το κεντρικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήπωτων δεν είναι σωστό αυτό της ΣΟΓΑΜΑ. Δηλαδή, η ΣΟΓΑΜΑ έχει λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ από τα Ταμεία Συνοχής έχοντας 51 της συνο συμμετοχή της ε, περιφέρειας της Γαλλικίας και 49% της υπηρεσίας αερίου. Ε, ε, το θέμα είναι ότι εδώ ε, θέλαμε τότε έπρεπε να σταματήσουν οι παράνομες χωματερές. Όμως η παρούσα κατάσταση έχει ως εξής η ισογάμα κάθε μέρα με φορτηγά ρίχνει ε, ε, χωρίς κανένα διαχωρισμό σκουπίδια και απόβλητα. Εδώ σας δείχνω φωτογραφία με τέτοια φορτηγά τα οποία ρίχνουν ε, τόνους ολόκληρους από απόβλητα χωρίς κανένα διαχωρισμό και χωρίς καμία ιεράρχηση. Ε, δημιουργούν αυτά τα, αυτές οι καταστάσεις μεγάλα προβλήματα στην γεωργία. Ε, η ε, ΣΟΓΑΜΑ δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις και δεν συμμορφούνται με τις οδηγίες και δεν είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο η Κομισιόν και να κρυφτεί πίσω από το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο καλύπτονται οι στόχοι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων ε, και ε, επίσης να απαγορευθούν παλιά ε, Thank Παλιά λατομεία να μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές. Ευχαριστώ επόμενος ομιλητής. οι πληροφορίες ε, που έχουμε εμείς ε, ε, είναι παρόμοιες με αυτές που μας έδωσε η Κομισιόν. Να πούμε λοιπόν και εξ ονόματος του ΕΛΚΟ ότι έχουν καλυφθεί όλες οι διαδικασίες αποτέφρωσης αλλά και αποφυγής πυρκαγιών. Επίσης γίνεται σεβαστή η ιεράρχηση των αποβλήτων. Υπάρχει ε, σχέδιο διαχείρισης ε, ε, αποβλήτων και γίνεται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση βάσει της αρχής ομολύνων πληρώνει. Επίσης ε, συμμορφούνται όλες οι διαδικασίες με την κείμενη νομοθεσία ε, και ε, οι εκπομπές είναι πολύ πιο χαμηλές από τις νόμιμες τιμές. Επομένως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες υπάρχει επομένως καλύπτονται όλα αυτά τα οποία καλύπτουν και το δικό ονόμασα πεδίο ε, δράσης. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αυτή η αναφορά γιατί κατανοούμε ότι πρόκειται για μια εσωτερική μάχη ε, στην Γαλλικία αλλά δεν χρειάζεται αυτή η εσωτερική μάχη να μεταφερθεί και εδώ. Η κυρία Μιράντα, 30 δευτερόλεπτα. Όχι, ε, ούτε η αρχή της, ε, ούτε συμμορφούνται με τις αρχές, ε, ούτε και με τις ενεργειακές εκπομπές. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν όλα σε αποτέφρωση. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει συμμόρφωση με την σχετική οδηγία. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία Έχουμε τα στοιχεία αξιολόγησης ε, ε, για το 2017. Ήδη το 2017 δεν υπήρχε ικανή συμμόρφωση, πόσο μάλλον το 2018. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η οδηγία, ε, συγγνώμη, αυτή η αναφορά, έτσι ώστε να μελετηθούν προσεκτικά τα στοιχεία του 2017. Ε, και επίσης ε, η χώρα μου δεν είναι περιφέρεια κυρία Εσταράσε και έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για, την, ε, για τα στερεά απόβλητα και τη διαχείρισή τους. Ωραία, είναι μερικοί που θέλουν να μείνει ανοιχτή, άλλοι να κλείσει. Έχω απαρτία, επομενω ψηφίζουμε. Ανοιχτή, ποιο θέλει να μείνει ανοιχτή, η γκουε και η πράσινη. Ποιος θέλει να κλείσει αυτή η αναφορά το ΕΛΚ και... Κοιτάξτε, θα πρέπει να ψηφίσετε, να σηκώσετε τα χέρια σα όσοι θέλετε να ψηφίσετε. Ωραία. Ξαναψηφίζουμε. Ποιο θέλει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Μετράμε λοιπόν. Ποιο θέλει να κλείσει αυτή η αναφορά. Ποιος απέχει. Δύο. Τρεις αποχές. Πέντε ε, υπέρ ε, του να κλείσει η ε, αναφορά. Άρα κλείνει η αναφορά αυτή. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη. Δεν είναι ε, παρόν ο αναφέρον. Επομένως πάμε στο σημείο 9. Πρόκειται για την αναφορά 0803. Πρόεδρος, να αφήσουμε τη συζήτηση για το προηγούμενο θέμα. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Ναι, έχουμε απαρτία. Έχουμε απαρτία. Είμαστε 12. Προχωρούμε λοιπόν. Επόμενο θέμα. Αναφορά 0803. ζητώ να προσπαθήσετε, ζητώ από όλους να προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν στις εργασίες της Επιτροπής μας. Για την αναφορά αυτή θέλετε το λόγο, κυρία Μιράντα. Διαδικαστικό. Ναι, αλλά να είναι πραγματικά διαδικαστικό. Σύμφωνα με, ποιον, με ποιο άρθρο. Okay, go ahead, but quickly. Εντάξει, σας δίνω το λόγο, αλλά γρήγορα παρακαλώ. Νομίζω ότι περίμεναν πέντε χρόνια οι αναφερόμενοι για αυτήν την αναφορά. Τέσσερα, τέσσερα χρόνια. Χρειάζονται λοιπόν να πάρω μια απάντηση. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να αφήσουμε ανοιχτή αυτήν την ε, αναφορά με τα νέα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι διαδικαστικό, λέει η Πρόεδρος. Αυτό δεν είναι διαδικαστικό. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι διαδικαστικό. Κοιτάξτε, οι κανόνες της δημοκρατίας ε, ε, αυτό επιτάσσουν. Καμιά φορά κερδίζει ένας, καμιά φορά κερδίζει ο άλλος. Αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά 0803. Είναι το σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως σχετικά με νέα βουλγαρική νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων και την σχετιζόμενη με αυτήν μη συμμόρφωση προς τα εφαρμοστέα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εν λόγω τομέα. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον, αλλά είναι εδώ εκπρόσωπος της Κομισιόν και του δίνω αμέσως το λόγο. Την 8 θα την κάνουμε μετά την αναφορά στο σημείο 8, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα ο ε, αναφέρον. Κομισιόν, παρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, ε, η αναφορά αυτή αφορά το νέο νόμο στη Βουλγαρία για τη διαχείριση των αποβλήτων που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Τροποποιήθηκε δε εκτοτέ επανειλημμένα πολλές φορές ε, για να ε, συμμορφωθεί απολύτως με την οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων. Μετά από την ε, σωστή, μάλλον επειδή η σωστή μεταφορά των οδηγιών είναι προτεραιότητα για μας, ο νέος νόμος αξιολογήθηκε αμέσως ως προς τη συμμόρφωσή του με την οδηγία πλαίσιο υπήρξαν στην αρχή κάποιες δυσλειτουργίες και αποκλήσεις, αλλά ακολούθησε γόνιμος διάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις βουλγαρικές αρχές, οπότε και τροποποιήθηκε ε, ως όφιλε η νομοθεσία αυτή και ε, μεταφέρθηκε σωστά στην βουλγαρική νομοθεσία η ελόγω οδηγία. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκλεισε τη διαδικασία αυτή πέρσι τον Οκτώβριο. Ε, οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Κανεί δεν θέλει το λόγο. Ε, ο κύριος Μαλίνοφ. Παίρνω το λόγο για να τα επιβεβαιώσω όλα αυτά. Ισχύουν. Η αναφορά ανάγεται στο 2011. Νομίζω ότι έπαιξε ένα θετικό ρόλο και για τα πρακτικά μόνο. Ε, δεν θυμάμαι να έχω ξαναζητήσει να κλείσει αναφορά, το ζητώ για πρώτη φορά. Μάλιστα, και εμείς το ίδιο λέμε να λάβουμε υπόψη ε, την πολύ σημαντική δουλειά και την πολύ ποιοτική που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέληξε ε, στην τροποποίηση της νομοθεσίας ε, της Βολερικής για τη διαχείριση των αποβλήτων και έκλεισε τον Οκτώβριο του 2017 το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Έχει οριμάσει η κατάσταση για να κλείσουμε την αναφορά. Πάρα πολύ καλή ε, αίσθηση της κατάστασης. Ωραία, δεν έχουμε για την 8 ακόμα τους αναφέροντες. Πάμε στο σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη που είναι αναφορά 1408 σχετικά με τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία όσον αφορά σχεδιαζόμενους χώρους υγειονομικής ταφής στο Δήμο Μοντάνα της Βουλγαρίας. Το όνομά σας δεν είναι εύκολο. Η κυρία ε, Αντωνέτα Ρίζοβα Καλάπης. Ε, σωστά το είπατε, έχετε το λόγο. Αυτή η αναφορά ε, έχει ε, τρεις αξιώσεις και καταγγελίες. Πρώτον, για τη διαχείριση της χωματερής στην πόλη Μοντάνα. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εξτάσει το θέμα αυτό και δεν κατέληξαν στην παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, γι' αυτό και έκλεισε το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Η δεύτερη αξίωση της αναφοράς ή ισχυρισμός ε, αφορά τις διαδικασίες που ακολούθησαν τα αρμόδια νομοθετικά και δικαστικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε, δεν είναι αρμόδια να επεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Ε, και ο τρίτος ισχυρισμός αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι εξέτασε τις ενδεχόμενες παραβιάσεις των απαιτήσεων ε, για πρόσβαση στη δικαιοσύνη των πολιτών σε ό,τι αφορά το, τις γενικές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις, τα κτίρια και ε, τους χώρους γενικότερα ε, υγειονομικής ταφής. Σε περίπτωση που καταλήξουμε ότι υπάρχει παραβίαση τη δομοθεσίας, νομοθεσία. θα αρχίσουμε ε, μια διαδικασία επί παραβάση προσφυγή. Αλλά αυτή η έρευνα δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη αναφορά. Έχει να κάνει με γενικότερα θέματα. Οι συνάδελφοι, ποιο θέλει το λόγο, ο κύριος Μαλίνοφ. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι την αναφορά κατέθεσε το Εθνικό Κίνημα Ecoglasnost που είναι το πρώτο περιβαλλοντικό κίνημα οικολογικό στη Βουλγαρία. Είχε ξεκινήσει ακόμα πριν την πτώση του κομμουνισμού. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστη οργάνωση αυτή και τα μέλη της ε, έχουν αποδείξει στην πράξη ε, την αποτελεσματικότητά τους. Είναι πολύ δίκαια η οργάνωση και πολύ ε, δραστήρια. Εγώ είμαι σε επαφή με τον αναφέροντα. Του επέστησα την προσοχή στο γεγονό ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μόλις μας παρουσίασε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απάντησή τους ήταν πολύ στεναρή ότι ακόμα δεν έχουν πρόσβαση και τους συμπεριφέρονται με τρόπο όχι σύνομο. Ε, με βάση την νομοθεσία που μόλις είπαμε ότι είναι καλή και μάλιστα εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι η αναφορά είναι πολύ παλιά. και με διάλογο μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Μπορούμε να την κρατήσουμε ανοιχτή, την αναφορά, έτσι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ε, ο αναφερόμενος να μας δώσει νέες προφορίες. Δεν ξέρω τα διαδικαστικά πόσο είναι τρει μήνες ή έξι και σε αντίθετη περίπτωση να την κλείσουμε. Και καλό θα ήταν να στέλνουμε και επιστολή στην περιφερειακή επιθεώρηση περιβάλλοντος και υδάτων, που είναι η αρμόδια υπουργική αρχή, για να τους ενημερώσουμε ότι οι Βούλγαροι πολίτες διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν πρόσβαση ε, ε, σύμφωνα με τον νόμο. Άρα, αν τους απαγορεύουν να πάνε, αυξάνονται οι υποψίες τους. Για να στείλουμε, λοιπόν, ε, στο τοπικό παραρτήμα του Υπουργείου αυτή την επιστολή και να αφήσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μας δώσουν νέα στοιχεία και μετά να κλείσει. Νομίζω έξι μήνες είναι μια πολύ λογική περίοδος. Αν αποφασίσετε όμως ε, διαφορετικά θα το δεχτώ και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το εξή. Συμφωνώ κύριε Μαλίνοφ, να την αφήσουμε ανοιχτή και να περιμένουμε ε, γραπτή ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιλωτική ε, διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό μόνο το λόγο θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν την πιλωτική έρευνα και να στείλουμε και επιστολή στις περιφερειακές αρχές λέγοντας ότι δεν το παρακολουθεί αυτό μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς όλοι στο θεσμικό μας όργανο και πολύ στενά μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Καλώς. Παραμένει απόν ο αναφέρον του σημείου 8. we are ending up in a very difficult situation. Τώρα έχουμε μπλέξει άσχημα. Το σημείο 8 είναι μια βουλγαρική, όχι διορθώνει, η ρουμανική αναφορά και μάλλον έχει χαθεί στις Βρυξέλλες ο Ρουμάνος αναφέρον κάτι το έχει συμβεί, δεν ξέρω. Δεν έχει φτάσει, δεν έχει χαθεί στο κτίριο. Α, κάπου στο δρόμο στις Βρυξέλλες. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται ή αποφάσισε να πάρει την επόμενη πτήση και να γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω, μυστήριο. Δεν σηκώνει και το τηλέφωνό του. Αυτό είναι το 8. Και ενώ το επόμενο θέμα, που είναι το 11, αναφορά 1569, η κυρία Μόια είναι αναφέρουσα, η οποία επίσης απουσιάζει και δεν έχει καταφτάσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχετε να πείτε κανένα θέμα έτσι δημοσίου ενδιαφέροντος ή ανθρωπίνου ενδιαφέροντος. Όχι. Why don't we take a pause of minutes? Να κάνουμε ένα διαλυματάκι 5-10 λεπτά. 10 και να δούμε αν θα έρθει κανείς. Ξαναρχίζουμε στις 11 και 4. You can always call your mom. They are always... Πάρτε τη μαμά σας τηλέφωνο. Χαίρονται οι μαμάδες όταν τις παίρνετε συνήθως. Πάντα έχετε συνήθως. Or your child. Ή το παιδί σας. Or have a quick coffee. Ή πιείτε κανένα καφεδάκι, εν πάση περιπτώσει, ραντεβού στις 11 και 4 και σε ελπίσουμε ότι θα έχουμε βρει μέχρι τον αναφέρον. Δεν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

Now we can restart the meeting. I think it's everyone should be here in just a matter of seconds. I already have a couple of... Ας ξαναρχίσουμε τη συνεδρίαση. Νομίζω πως σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι όλοι εδώ. Ε, ζητώ συγγνώμη για το πώς έγιναν όλα. Ξέρω πως η κυρία Γιολάντα Μόγε βρίσκεται εδώ και με χαρά σας καλωσορίζω στην Επιτροπή για την 1569 ε, πολεοδομικό σχέδιο για ε, μια μολυσμένη τοποθεσία στην πόλη του Λουξεμβούργου. Oui, mais le micro, s'il vous plaît. Oh, pas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 Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα μετά από δύο χρόνια και λίγους μήνες μετά από την υποβολή αυτής της αναφοράς η απορρίπανση αυτού του χώρου έχει περάσει τις πιο ε, επικίνδυνες φάσεις. Τώρα είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο όλων αυτών των εργασιών που έχουν ήδη γίνει. Όμως μια εξωτερική και ανεξάρτητη ε, έρευνα θα μας βοηθήσει για να μας καθησυχάσει μέχρι στο τέλος το του project. Επίσης θέλαμε η υγεία των ε, περίοικων να, να αναλυφθεί από το Λουξεμβούργο και την κυβέρνησή του. Γι' αυτό ήρθα εδώ ε, να υπερασπιστώ αυτό το κείμενο στο όνομα των ε, ε, γειτόνων μου ε, στο γειτονιά αυτή του Λουξεμβούργου. Από το 2017 η επικοινωνία και η διαφάνεια της πόλης του Λουξεμβούργου και της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου βελτιώθηκε πολύ. Η στάση τους είναι πολύ πιο θετική και συνεργαστική. Και τώρα θα προχωρήσω με τα γιατί με τους λόγους για τους οποίους κάναμε αυτή την αναφορά. Το 2015 είδαμε πως είχε εγκριθεί ένα ε, project ε, για την κατασκευή ε, ε, κτηρίων στο, στο, στη δική μας περιοχή που ήταν πολύ μολυσμένη με διάφορα υδρο, υδρογονάνθρακες ε, και διάφορες καρκινογόνες ουσίες για... είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες για την ανθρώπινη υγεία. Ε, Ξατμίζονται δε πολύ εύκολα στον αέρα και μπορούν να συμπυκνωθούν εκ νέου και να ε, εισχωρήσουν στο έδαφος και στο νερό κατά τη διάρκεια της ε, ε, επεξεργασίας αποβλήτων παράγονται ή μέσω της αποθήκευσης ή μέσω του συστήματος ποιόσιμου νερού. Σημαίνει πως το αναπνέουμε, το πίνουμε, τις πίνουμε και ότι βρίσκονται στους στίχους μέσα κτηρίων που ε, βρίσκονται κοντά σε αυτή τη ρυπασμένη, ε, μολυσμένη περιοχή. Είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό και κάθε μία από τις μολύνσεις αυτές έγιναν ανάμεσα στα έτη 2001 και 2003. Η πόλη του Λουξεμβούργου γνώριζε ήδη την τοξικότητα αυτών των ουσιών από το 1998, ωστόσο η δήμαρχος Πολβά, που είναι και σήμερα δήμαρχος της περιοχής, το 1999 συνεννοήθηκε με έναν από τους ιδιοκτήτες της βιομηχανικής ζώνης και ξεκίνησε ε, συζητήσεις ε, που ε, ολοκληρώθηκαν το 2000 και τελικά δόθηκε η άδεια κατασκευής ε, ε, από την πόλη του Λουξεμβούργου από τον κύριο Μπέρμικε που, είναι που ήταν τότε ο δήμαρχος της πόλης και αυτό χωρίς εξυγίανση της περιοχής. Ε, εν τω μεταξύ οι περίοικοι έχουν προβλήματα μνήμης, ε, ε, αναπνοής, δύσπνιες και το πρόβλημα του πόσιμου νερού ε, σημειώθηκε από εδώ και καιρό ήταν ένας πολύ μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε και το 2014 ο κύριος Κορτσέλη διοκτήτης ε, ε, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ποινικά. Ένα χρόνο μετά, ο κύριος Κορτέρη πούλησε την ιδιοκτησία του στην Όμιλο Αλφίν, του οποία ο κύριος Πολ Χέλμιγκερ, πρώην δήμαρχος του Λουξεμβούργου, ήταν στο, συμβούλιο, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο το Δημοτικό Συμβούλιο με την κυρία Λιδή Πόλβα ως ε, δήμαρχο αυτή τη φορά εγκρίνει την ε, ε, ανάπτυξη αυτής της ζώνης κατοικιών και γραφείων από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η απορρίπανση, ο καθαρισμός, η εξηγήση του χώρου. Φυσικά οι γείτονε ε, συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Έχουν στείλει εκατοντάδε επιστολέ διαμαρτυρία στην ε, Δήμαρχο και στην Υπουργό Περιβάλλοντο. Ακόμα και ο διαμεσολαβητή έστειλε δύο ε, επιστολέ αρχέ 16 και μέσα 17 στην Δήμαρχο Πολφά. Κανεί δεν έχει πάρει απάντηση. Εν τω μεταξύ φτιάξαμε αυτή την αναφορά τον Απρίλιο του 2016. Τον Άνοιξη του 2017 είχαν ήδη αρχίσει οι εργασίες και μαζί τους και οι παρατυπίες. Καμία ενημέρωση, καμία διαφάνεια, καμία απάντηση στα αιτήματά μας. Άνθρωποι που διαμαρτύρονταν για ε, την σκόνη και τη μόνιμη ε, ε, τη βρωμιά που προερχόταν από αυτό το εργοτάξιο και επειδή οι εργάτες δεν έβρεχαν το χώρο στη διάρκεια των εργασιών. Ε, ο τύπος ήρθε στις 30 Ιουνίου 2017. Ο κ. Μάρκ Άγγελ, που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε επίγουσα ερώτηση στην κυρία Πόλβα για την έλλειψη διαφάνειας και επικοινωνίας για ε, το project Paul ε, Δήλωσε πως δεν είχε γίνει καμία καταγγελία για αυτό το project τότε και ότι δεν υπήρχε ούτε διαφάνεια ούτε επικοινωνία γιατί δεν υπήρχαν απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, το 4 Ιουλίου 2017, ο βουλευτής ε, Σελος μίσμε, έθεσε μια, μια ερώτηση που αφορούσε τον έλεγχο της ρήπασης του χώρου και των υδάτων καθώς και τα προληπτικά μέτρα και τα επιοπτικά μέτρα που είχαν ληφθεί για την προστασία εργαζομένων και περίοικων. Κοινή απάντηση της Υπουργού Περιβάλλοντος και Υπουργού Εργασίας έφτασε το Σεπτέμβριο και ήταν εντυπωσιακή ότι δηλαδή η υγεία των περιοίκων δεν ήταν δική τους ευθύνη. Ε, τότε εμείς όλοι οι περίκοι θήκαμε ότι είχαμε μπει στην άκρη και ότι ήμασταν τελείως αδύναμοι. Τώρα έχετε όλα τα στοιχεία που τα 5-7 λεπτά μου επέτρεψαν να σας δώσω. Σας ευχαριστώ και δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Όπως και στην προηγούμενη αναφορά στην οποία αναφέρθηκα, υπάρχουν κάποια στοιχεία αρχής. Εδώ έχουμε βεβαίως μία μεμονωμένη ε, ε, περίπτωση ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατανοεί βεβαίως ε, τον προβληματισμό ε, που σχετίζεται με την υγεία των αναφερομένων. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι σε τούτη την συγκεκριμένη περίπτωση ε, μπορεί να υπάρξει κάποια Ε, μπορεί να υπάρχει παρατυπία, αλλά θα πρέπει αυτή ε, και μη συμμόρφωση, αλλά θα πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί από τις εθνικές αρχές. Ε, αυτές μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από την Κομισιόν στο να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επομένως, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από την αναφορά ε, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει σαφής παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Η ε, αναφερόμενη δεν φαίνεται να ε, καταδεικνύει διαρθρωτικό πρόβλημα και επομένως η Κομισιόν δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτήν την αναφορά. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θέλουν οι συνάδελφοι μήπως να πάρουν το λόγο. Όχι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σαφής περίπτωση δεν φαίνεται να καταδεικνύεται διαρθρωτικό πρόβλημα το οποίο να σχετίζεται με την μη εφαρμογή ε, του ε, ενωσιακού νόμου. Η Κομισιόν έχει την άποψη ότι ε, πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση του θέματος είναι οι εθνικές αρχές και νομίζω ότι και για και ε, από ό,τι καταλάβαμε και από την ίδια την ε, αναφέρουσα, ε, έχει βελτιωθεί η συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και το Υπουργείο και επομένως εγώ προτείνω να κλείσει αυτή η αναφορά. Συμφωνείτε όλοι, πολύ ωραία, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε... is the, the first να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως. Ε, πρόκειται για την αναφορά 0581 σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά τη συλλογή και αποτέφρωση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ε, στο έδαφος της Ρουμανίας. Α, έχασε το αεροπλάνο ο, ο αναφέρον και επομένω δεν είναι καθόλου στις Βρυξέλλε. Έχει μείνει στη Ρουμανία γιατί έχασε το αεροπλάνο. Επομένως δεν θα του δώσουμε το λόγο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της αναφοράς αυτής. Έχουμε τον κύριο Ντίας Δελκαστήγιο. Ε, παρακαλώ διαφωτίστε μας σχετικά με την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς εδώ διαπιστώνουμε δύο σημεία. Πρώτον, σύμφωνα με, τη, τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, οι ρουμανικές αρχές έχουν ε, πάρει τα απαραίτητα μέτρα ε, έτσι ώστε να ε, μην υπάρξουν επικίνδυνες εκπομπές από την αποτέφρωση ιατρικών αποβλήτων. Δεύτερον, ο αναφέρον αναφέρεται σε μαφιόζικες ε, διεργασίες ε, και σε απο... φοροδιαφυγή από την ε, αρμόδια εταιρεία. Η Κομισιόν δεν έχει άμεση αρμοδιότητα για τέτοια θέματα. Αυτά θα πρέπει οι αρμόδιες εθνικές αρχές να τα αντιμετωπίσουν. Ως γενικό κανόνα, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ε, άμεση ευθύνη για την σωστή εφαρμογή ε, και ενσωμάτωση της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Κομισιόν πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές ορθώς εφάρμοσαν την νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ο αναφέρον πάντως μας έστειλε κάποιες ε, τελευταίες φωτογραφίες σχετικά με επικίνδυνη ιατρικά απόβλητα. Πρέπει να πούμε ότι στην ε, Ρουμανία ε, καλύφθηκε επικοινωνιακά πολύ το θέμα αυτό και πρόκειται πάντως για μια κατάσταση όπου η Κομισιόν δεν μπορεί να λέει ότι οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, αυτό μας είπατε. Οι επιθεωρήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα μάλλον να το πούμε διαφορετικά, έγιναν κάποιες επιθεωρήσεις και ο ίδιος αναφέρει ότι δεν, έγινε, δεν ελήφθησαν υπόψη ε, γνωστές και τεκμηριωμένες παραβιάσεις από την πλευρά ε, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ε, ε, αποτέφρωση αυτών των, των ιατρικών αποβλήτων. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αν θέλετε να κλείσει η αναφορά, παρακαλώ να μου το πείτε. Okay, if, if nobody... Jude. Jude. Απόψη μου είναι ότι ε, μια και είχε ένα πρόβλημα ο αναφέρον και δεν ήταν ότι δεν ήθελε να έρθει, ίσως καλό θα ήταν ε, πρώτα να ελέγξουμε αν έχει επικαιροποιημένες ε, ε, πληροφορίες και ίσως οι συντονιστές να αποφασίσουν τι θα γίνει με αυτή την αναφορά, αν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς περιμέναμε να ακούσουμε τα σχετικά από τον ε, αναφέροντα και δεν έχουμε και κανένα Ρουμάνο συνάδελφο εδώ παρόντα και επομένως ε, είναι λίγο δύσκολο να κρίνουμε μόνοι μας. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Ε, νομίζω ότι καλύτερα να δώσουμε φωνή ας πούμε στον αναφέροντα που δεν είναι εδώ και εγώ την ίδια άποψη έχω. Από τη μια μεριά λέω ωραία δεν ενδιαφέρθηκε αρκετά έτσι ώστε να έρθει έγκαιρα εδώ ε, ο αναφέρον αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ας σκύψουμε λίγο πάνω από το θέμα αυτό να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά να στείλουμε ε, μία επιστολή στις αρμόδιες ρωμανικές αρχές έτσι ώστε να έχουμε και τη δική τους άποψη γιατί από ό,τι καταγγέλει ο αναφέρον ε, συνεχίζονται οι παρανομίες εκεί ε, ενώ η Κομισιόν μας λέει ότι δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε το θέμα ανοιχτό και να κοινοποιήσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ενδιαφερόμαστε για το θέμα και το κρατάμε ανοιχτό. Ωραία, λοιπόν, έτσι θα κάνουμε. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την θέση σας. Ωραία, ολοκληρώθηκαν οι πρωινέ εργασίε. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30 το απόγευμα. Όχι ακριβώ, δηλαδή. Ε, θα πάμε στην κοινή συνεδρίαση ε, στην, ε, στην αίθουσα 5Β001. Δηλαδή θα μπείτε στο σανσέρ και θα πατήσετε το κουμπί 5. And the meeting starts at 11.50, so it gives you 18 minutes. 11 και 50 θα ξεκινήσει αυτή η κοινή συνεδρίαση. Έχετε λίγο χρόνο λοιπόν μέχρι να καταφέρετε να βρείτε την αίθουσα.